So, dear colleagues, uh, the uh, Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρία της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, χωρίς τις γυναίκες. Ε, είναι σκέτη η Επιτροπή μας, ε, πολύ λίγοι παρόντες οι βουλευτές. Θα δώσω μέσα το λόγο στον Ερίκο Γκασπαρά. Ευχαριστώ θα είμαι πολύ, πολύ συνθετικός, δεν θα τα πω πολύ απλά, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για το θέμα. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε γνωμοδότηση για το θέμα το οποίο, μας έχει, το οποίο επιβλήθη την 10η Δεκεμβρίου από τον ε, Πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης και θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε ε, μέχρι την 17η Νοεμβρίου και Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε στις 3 Δεκεμβρίου τη συζήτηση στην ε, Αρμόδια Επιτροπή. Πρόεδρος, μπορώ να ζητήσω ησυχία και να ζητήσω από όσους δεν ενδιαφέρονται για το θέμα να εγκαταλείψουν ησύχως την αίθουσα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ή στις 15 Δεκεμβρίου έτσι ώστε να έχουμε την ε, δυνατότητα να γνωρίσουμε όλοι ε, το θέμα γιατί δεν το ξέρουμε ακόμα ακριβώς. Το θέμα βεβαίως είναι πολύ ενδιαφέρον αλλά είναι περίπλοκο ταυτοχρόνως και οπωσδήποτε είναι ένα ε, ζήτημα το οποίο ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να, να το μελετήσουμε προσεκτικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια έχει εκπονήσει 30 περίπου νομοθετήματα, αλλά το θέμα είναι περίπλοκο και ε, έχει τόσες ε, πολλές πτυχές που δεν μπορούμε να φανταστούμε βεβαίως πλήρη εναρμόνιση για όλες τις χώρες μέλη. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την νομοθετική ε, διαδικασία που έχει ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που έχουν λάβει 18 χώρες της είχαν λάβει 18 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορούμε να σκεφτούμε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα ελάχιστα πρότυπα, τα minimal standards έτσι ώστε να γίνει αποδεκτή μια πρόταση από όλους. Μου ζητήθηκε να είμαι σύντομος, ήμουν σύντομος, ευελπιστώ ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία με τους συναδέλφους έτσι ώστε να ε, εκπονηθεί και μια καλή γνωμοδότηση. Είμαι στην διάθεση των συναδέλφων έτσι ώστε ε, μέχρι τη 17η να ε, ε, έρθουν σε επαφή μαζί μου οι συνάδελφοι αν θέλουν να μου υποβάλουν κάποιες σκέψεις. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκασμπάρα. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο για την παρουσίαση. Το θέμα είναι πολύπλοκο, ξεκινώντας ήδη από την νομική βάση. Βλέπουμε πως εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε κάποιους κανονισμούς με τους οποίους επιβάλλουμε κάποια συμπεριφορά στα κράτη-μέλη και πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει διαβούλευση με τους εργαζόμενους, εκπροσώπηση. Εγώ στη χώρα μου έχουμε εμείς πάρα πολύ καλή εκπροσώπηση των εργαζομένων, αλλά όπως είπατε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να μην παραβιάσουμε την αρχή της επικουρικότητας και να μην εμποδίσουμε την δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος λόγο, όχι. Κύριε Κασφάρα, καλή τύχη. Περνάμε στο επόμενο θέμα λοιπόν. Πρόσβαση στα έγγραφα, η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω πως είναι πέμπτη απόγευμα. Δεν θα δείξω λοιπόν το, θέμα, το πάθος μου για το θέμα. Λοιπόν, αποφασίστηκε πως η Επιτροπή μας θα πρέπει να γνωμοδοτήσει προς την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την εφαρμογή του κανονισμού για την πρόσβαση στα έγγραφα Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιών. Το λεγόμενο 1049 του 2001 που είναι η πρόσβαση στα έγγραφα και την χάνει ο εισηγητής ή η εισηγήτρια να είναι και μέλος και της δικής μας επιτροπής και να είναι και στη Λίμπε η κυρία Φερέρα. Ελπίζω λοιπόν να συνεργαστούμε για να δούμε πώς η επιτροπή μας μπορεί να στηρίξει την έκθεση αυτή στη Λίμπε. Να τονίσω την σημασία κάποιων πρόσφατων αποφάσεων του ΔΕΚ που λένε πως τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να τα παίρνουμε σοβαρά σε κάθε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναφέρω μόνο τα όσα αναφέρονται στην απόφαση περί ψηφιακής ε, απομόνωσης. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα πάντα βεβαίω εντό των πλαισίων. Τώρα, τα δεν μπορούμε να τα γράψουμε όλα, αλλά... Θεωρώ πως θα πρέπει να δούμε κάποια βασικά ζητήματα και κάποιες πρόσφατες αποφάσεις. Ε, τα τρία ζητήματα λοιπόν αυτά είναι πρώτον πρέπει να υπενθυμίζουμε στα θεσμικά όργανα τα διοικητικά τους καθήκοντα γιατί κανένας πολίτης δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του για πρόσβαση στα έγγραφα ε, εκτός εάν η διοίκηση είναι οργανωμένη και κρατάει αρχεία. Να επισημάνω πως από καιρού καιρών φαίνεται πως υπάρχει ξανά μια νέα κατηγορία εγγράφων που δεν μπαίνει στα αρχεία που απαιτεί ο κανονισμός αυτός. Οπότε με το να επιμένουμε στο καθήκον της διοίκησης να τηρεί αρχεία νομίζω πως μπορούμε να φωτίσουμε και κάποιες σκοτεινές πτυχές της δραστηριότητας της Ένωσης που θα έπρεπε να γνωρίζουν οι πολίτες. Υπάρχει επίσης μια άλλη σύμπτωση που αφορά τον κανονισμό ε, για τις διοικητικές διαδικασίες και υπάρχει ένα προτινόμενο άρθρο που αφορά ακριβώς ε, την τήρηση αρχείων. Υπάρχει λοιπόν, όπως είπαμε, η οργάνωση των πληροφοριών που είναι προαπαιτούμενο. Μετά, κατόπιν, πρέπει να δούμε κάποιες συνταγματικές πτυχές ε, που έχουν ενισχύσει την πρόσβαση του κοινού, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις την περιορίζουν. Και νομίζω πως ε, Είχαμε και αυτή τη συζήτηση σήμερα το πρωί με τον κύριο Φερχώστα για την καλύτερη νομοθεσία και στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαμε να δούμε ε, πώς ε, κολλάει αυτό με το δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση στα έγγραφα. Και βέβαια αντιλαμβάνομαι πως το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή για το Κοινοβούλιο είναι να έχουμε εμείς πρόσβαση στα έγγραφα του Συμβουλίου για να ξέρουμε το τι κάνει ο συνομοθέτης. Και αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Αλλά υπάρχει μια άλλη διάσταση, βαθύτερη, που αφορά το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών και με την άδειά σας ε, θα το εξετάσω αυτό και θα κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις. Τρίτον, θα ήθελα να κοιτάξω τις ελλείψεις ε, των θεσμικών οργάνων και την αποτυχία τους στην εφαρμογή των αποφάσεων του Κοινοβουλίου. Το κοιτάμε ακόμα, αλλά θα πρέπει να δούμε το, εμείς το τι δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Και ακριβώς αυτό είναι το θέμα, το πεδίο εφαρμογή της ε, γνωμοδότησης, το οποίο είναι η εφαρμογή του υφιστάμενου κανονισμού. Και θα ήθελα εδώ πέρα να δω πώς η διοίκηση του Κοινοβουλίου αντιμετωπίζει τα αιτήματα του κοινού για πρόσβαση στα έγγραφα, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν κάνουμε, δεν τηρούμε τα όσα λέμε. Εγώ και χάρη σκέφτομαι εδώ πέρα κάποιες αποφάσεις ε, του Προεδρείου του Κοινοβουλίου και κάποια γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία. Λοιπόν, καλό θα ήταν να έχουμε μια σύντομη γνωμοδότηση. βεβαίω η κυρία Φερέρα κάνει πολύ πιο εκτεταμένη δουλειά και τελευταία πρόταση είχα συντάξει τη σχετική έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ το 2011 και τότε σχεδόν ομόφωνα το 2011 είχαμε πει κάποια πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν γίνει. Thank you, uh, Madam Hautala. Ευχαριστούμε κυρία Χαουτάλα. Δεν ε, βλέπω να ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Νομίζω ότι όλα αυτά που μας είπατε ε, είναι εξαιρετικά και συμφωνούμε απόλυτα με τον τρόπο τον οποίο θέλετε να προχωρήσετε. Πρέπει να πω κάτι για το 20. Ο κύριος Χρυσόγονος δεν είναι εδώ, αλλά πρέπει να σας πω ότι ε, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 19η Νοεμβρίου και επίσης είναι σημαντικό να πω ότι θα πρέπει να γίνουν οι τροπολογίες να γίνουν επί της εκθέσεως και όχι επί του μνημονίου συνεργασίας. Ε, μόνο την έκθεση μπορούμε να τροποποιήσουμε, να υποβάλουμε τροπολογίες δηλαδή. Τελευταίο σημείο Η επόμενη συνάντη, συνεδρίασή μας, Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου το απόγευμα και, συγγνώμη, το πρωί και το απόγευμα. Μέχρι δηλαδή τις 6.30 το απόγευμα. Βλέπετε ότι κάνουμε εντατικά μαθήματα προετοιμασίας για την Προεδρία. Ευχαριστώ. So, and I will... Thank you. I will disappear now. Thank you much. Okay.